Good morning, colleagues. Um, Καλημέρα σας, συνάδελφοι. Πάμε στο σημείο 1, η έγκριση της ημερής διάταξης. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ, καθίστε. Γλωσσικό προφίλ, συνάδελφοι. Σημειώστε ότι έχουμε διερμηνία από γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ε, ολλανδικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ε, ουγγρικά και τα λοιπά. Είστε έτοιμοι, παρακαλώ να ελέγξω συνάδελφοι. Ξέρω, Μόνικα, εσύ είσαι πάντοτε ετοιμοπόλεμη. Το ξέρω, αλλά οι υπόλοιποι. Να ελέγξουμε γιατί εδώ έχουμε μόνο ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Μήπως κανείς δεν έχει φέρει την κάρτα του να μας το πει. Ένας το έχει πει, θα καταγραφεί η ψήφος του, άλλος κανείς. Σεσίλια, και εσύ ξέχασες την κάρτα σου. Αγαπητέ Κλοντ, μας λες κανένα αστείο, μας λες κανένα τραγουδάκι, γιατί έρχεται η κάρτα μου. φιλελεύθεροι πραγματικά. Εντάξει, λοιπόν. Εδώ σας έχω ειδοποιήσει εδώ και εβδομάδες, Σεσίλια. Άντε, ας κάνουμε ένα διαλυματάκι, δύο λεφτά. I'm going to, uh, before we vote, I'm going to give the floor to each of the rapporteurs, so... Θα δώσω το λόγο στους εισηγητές. Ας αρχίσουμε μέχρι να καταφτάσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Τώρα έχετε όλη την ε, κάρτα ψηφοφορία σας. Ωραία, καθίστε. Συνάδελφοι, σημείο 4. Έχουμε την προστασία ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αρμόδιες αρχές με στόχους πρόληψης, έρευνας, ανείχνευσης, ιδίωξης ε, ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών ε, ποινών μάλλον ε, και την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων. Εισηγητής είναι ο κύριος Λαουριστίν. Μετά από το σχέδιο σύστασης για την οδηγία για την ε, προστασία των δεδομένων και την έναρξη της προθεσμίας για τις τροπολογίες δεν κατατέθηκα μία τροπολογία εντός του χρονικού ορίου και άρα σύμφωνα με το κανόνα κανονισμό 66 θα ψηφίσουμε άμεσα για το σχέδιο που υπέβαλε ο εισηγητής. Πριν να... Ε, η εισηγήτρια με συγχωρείτε. Κυρία Λορεστίν, θέλετε το λόγο σύντομα. Ναι, ευχαριστώ στο Κλοντ. Ε, θέλω θερμά να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, όλους τους σκιώδεις εισηγητές, όλους τους βοηθούς μας και τους εκπροσώπους της Κομισιόν και του Συμβουλίου, διότι ε, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά. Εδώ η οδηγία αυτή που αποκαλείται οδηγία για την αστυνομία ήταν πολύ δύσκολη. Υπήρξαν ένα σωρό αντιφατικές απόψεις και γνώμες ανάμεσα στους βουλευτές, ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες, ανάμεσα στους συναδέλφους Έγινε πολύ σκληρή δουλειά σε πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας, κάποιες φορές πολύ έντονες συζητήσεις, αλλά τελικά καταλήξαμε σε κοινέ λύσεις και τώρα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό ψηφίστηκε ήδη από την ε, δική μας ε, ομάδα και ελπίζω πως έτσι θα το ψηφιστεί, υπερψηφιστεί και εδώ και βεβαίως θα ψηφίσουμε και για την λύση όλων αυτών των προβλημάτων. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι αύριο θα αρχίσει η εφαρμογή. Ελπίζω πως όλοι μας θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στις χώρες μας αυτή τη διαδικασία, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε το νοοτροπία της επιβολής του νόμου σε όλες τις χώρες που θα περιλαμβάνει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, των ανθρώπων ως κομμάτι της καθημερινής δουλειάς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θέλουμε οπωσδήποτε να το πετύχουμε. Ευχαριστώ, Μάριο. Να προχωρήσουμε. Ας ε, προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 45 ψήφοι υπέρ προς 4 με μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. So, colleagues, we move now to the second vote. Δεύτερη ψηφοφορία τώρα. Προστασία των τόμων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων κανονισμός, ε, γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων. Μετά από την υποβολή του σχεδίου ε, ε, ψηφίσματος και την έναρξη της χρονικής προθεσμίας για υποβολή τροπολογιών δεν κατετέθη καμία τροπολογία οπότε σύμφωνα με το κανόνα 66 θα ψηφίσουμε κατευθείαν για το ψήφισμα που υπέβαλε ο εισηγητής ο κύριος Άλμπρεχτ που είναι εισηγητής είναι εδώ και θέλει να πάρει το λόγο σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, αν και τα περισσότερα υπόθηκαν εχθές στην παρουσίαση όπου ευχαριστήσα, ε, όπου μάλλον ευτυχώς η συνάδελφος Κέλλερ διάβασε τις δικές μου παρατηρήσεις. Εγώ θέλω να μοιραστώ τις ευχαριστίες για όλους όσους ασχολήθηκαν, προς όλους όσους ασχολήθηκαν και εργάστηκαν εντατικά ώστε να βρεθεί λύση και αποτέλεσμα για αυτό το πακέτο μεταρρύθμισης. Ήταν πολύ δουλειά για όλους. Πέντε χρόνια συζήτησης τουλάχιστον σε αυτό το κοινοβούλιο και για τον μεγάλο κανονισμό της προστασίας των δεδομένων ε, είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά για την ψηφιακή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά μόνο αυτό θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα για την περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο της ε, εφαρμογή του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των δεδομένων παντού στην ε, ενωμένη αγορά με ένα αρμονισμένο και συνεπή τρόπο, πράγμα που θεσπίζει προδιαγραφές και για μας τους Ευρωπαίους ώστε να προχωρήσουμε και να διαπραγματευτούμε σε περισ... για διεθνείς προδιαγραφές στον τομέα των ε, δεδομένων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι επί τη βάση ε, των όσων ισχύουν ως θεμελιώδης αξία και ήταν γι' αυτό πολύ σημαντικό το να φτάσουμε σε συνένεση. Είμαι ευτυχή που αν και προσπαθήσαμε να βρούμε την ισορροπία μέχρι την τελευταία στιγμή και από την αρχή ήταν πολύ έντονη προσπάθεια στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τελικά ποτέ δεν χάσαμε δεν ξεχάσαμε την ιδέα της εξέβρεσης ισορροπίας με όλους, έτσι ώστε αυτή η συμβιβαστική να, μπει σε, να δεθεί σε πράξη και να φτάσουμε σε μια θετική κατάσταση για τους ελεγκτές των στοιχείων καταρχάς που χρειάζονται νομική βεβαιότητα, αλλά και που και για τους καταναλωτές, τους πολίτες που χρειάζονται εμπιστοσύνη για την εφαρμογή του, του δικαιώματός τους, για την προστασία του των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και επιγραμμικά online. Τεράστια ε, λοιπόν προσπάθεια και η προσπάθεια της κυρίας Λορεστίν για την εφαρμογή και την πραγματική ε, υλοποίηση αυτού του νέου νομικού πλαισίου θα είναι πολύ θετική για την ενιαία αγορά Ελπίζω πως θα το δουν όλο αυτό σαν ευκαιρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η γραμματεία, και εγώ το βλέπω ως εισηγητής, η γραμματεία κάνει πολύ εντατική δουλειά, αν και πολύ συχνά γίνεται στα παρασκήνια. Πολύ συχνά μένει και δουλεύει ολονυχτίες. Ε, κάνει ολονυχτίες για να τελειώσουν όλες οι εργασίες. Θέλω να επενέσω τη γραμματεία που κάνει τεράστια προσπάθεια υπέρ της δημοκρατίας μας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Jan. Ευχαριστώ πολύ, Γιάν. Επειδή θα φύγουμε μετά την ψηφοφορία, να πω ότι αν υπερψηφίσετε θα είναι το τελευταίο κομμάτι του πακέτου της ΛΥΜΠΕ και στη συνέχεια θα υποβληθεί ε, στην Ολομέλεια για ψηφοφορία. Ένας ψηφοφορίας λοιπόν. The vote is closed. ψηφοφορίας with one abstention. Congratulations to the rapporteur. Thank you, colleagues. That's the end of voting time, and thank you for your patience. Ευχαριστούμε, Λέξη. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή στη συνεδρία της ΛΥΜΠΕ.